Pan Przewodniczący! Dzień dobry, proszę Państwa o zajęcie. Καλημέρα Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 7 kwietnia 2011. Και για τη συνεδρίαση που είχε διακοπεί συνεχίζεται με τη σημερινή μας συνεδρίαση τα πρακτικά του τη συνεδρίαση είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Και έτσι θεωρείται ότι κυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Κάποιες παρατηρήσεις για την έναξη της συνεδρίασης. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα στην Φλωρεντία και όπως γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έχει την έδρα του στην Φλωρεντία και το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ η Γιορτή της Ευρώπης διεξάγεται εκεί υπήρξε και μια συνεδρίαση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναντήθηκα και με φοιτητέ του Πανεπιστημίου είναι η 61η επέτειος της διακήρυξης του Ρομπέρ Σουμάν διακήρυξης που οδήγησε μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα. Θα ήταν περήφανο ο Ρόμπερ Σούμαν για αυτά τα οποία πετύχαμε. Οι πατέρες οι ιδρυτές γνώριζαν ότι οι κρίσει υπάρχουν για να τις ξεπερνάμε και ότι χρειαζόταν ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη, ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη. Γι' αυτό προσβλέπουμε με ελπίδες ε, προς το μέλλον σε αυτή τη συγκυρία. Επόμενη πληροφορία που θα ήθελα να σας δώσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα είναι πλέον πλήρες μέλος της, Ευρω... της ε, παγκόσμιας κοινότητας, της παγκόσμιας κοινότητας. Στις 3 Μαΐου τα Ηνωμένα Έθνη δέχθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό αυτό το καθεστώς και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να προσφωνήσει και να απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι επίτευγμα κοινό της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε με μία φωνή ενωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντική η δράση και η δραστηριοποίηση με σθένος σε αυτή τη συγκυρία διότι είναι μια χρονική συγκυρία που πρέπει να δράσουμε όλοι μας και να δρούμε και στην Βόρεια Αφρική και στη Συρία και στον Παχρέν όπου βλέπουμε κρίσεις να ξεδιπλώνονται μπροστά μας, εξεγέρσεις. Στις 17 Μαΐου θα γιορτάσουμε την επέτειο κατά της ομοφοβίας. Δυστυχώς παγκόσμια πρέπει να πούμε ότι διώκονται άνθρωποι και σκοτώνονται, δολοφονούνται ακόμα επειδή είναι ομοφιλόφιλοι. Στις συνθήκες και στην χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για να μπορέσει να ξεριζώσει, να εκριζώσει την ομοφοβία. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει, ούτως ή άλλως έχει καταδικάσει την θανατική ποινή που έχει επιβληθεί και επιβάλλεται σε άτομα από το, τις του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της συμφιλίωσης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Και τώρα περνάμε στην κανονική μας εργασία σύμφωνα με την ημερησία διάταξη και πρέπει να πω ότι από πλευράς Ντεπαλέστρης εθίγει ένα θέμα υπήρξε ένα αίτημα το οποίο επανελήφθηκε και του κυρίου Σπένσκι και του κυρίου Βάντιμ Τούντο. ζήτησαν να μπορέσουν να επωφεληθούν από το καθεστώς των κοινοβουλευτικών ασυλιών και θα απευθυνθούν τα αιτήματά τους στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Τούτων λεχθέντων διαδικαστικό εσείς παρακαλώ. 847 παρακαλώ. Δεν κατάφερα να κατανοήσω. Με ακούτε. Δεν κατάφερα να καταλάβω αυτά που είπατε. Ο κύριος Magistris ζήτησε, αν κατάλαβα καλά, να μην αρθεί η ασυλία του. Τι είπατε. Κοιτάξτε, ο κύριος Ντεματζίστρης ε, στην χώρα μου είναι ο πρωταθλητής εναντίον της διατήρησης της ε, ασυλίας. Οπότε ίσως να υπάρχει εδώ ένα λάθος στη μεταφορά του νοήματος. Παρακαλώ να διευκρινίσετε αυτό το οποίο είπατε για τον κύριο Ντεματζίστρης. Yes,